Bene, allora possiamo cominciare. Anche perché Καλημέρα σας. Ας αρχίσουμε παρακαλώ, γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες και θέλω να τις ξεκινήσουμε στην ώρα, στην ώρα τους. Παρόλο που δεν έχουμε πολλούς παρόντες, αλλά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι εδώ. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για το θέμα αυτό θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κρόιτσμαν. Ja, vielen Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ τους ε, συνεισηγητές, τους σκιώδησηγητές και τους λοιπούς συναδέλφους που έχουν συμβάλει. Οι περισσότερες τροπολογίες. On... Τίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα του προπολογισμού, της ε, επικάλυψης μέτρων, κυρίως και Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε κυρίως ε, εισαγάγει στην ε, πρότασή μας. Προσπαθούμε για να έχουμε ένα κείμενο σχετικά ισχνό και ευνόητο να ε, έχουμε, θα αναγκαστούμε λοιπόν να διαγράψουμε κάποιες τροπολογίες, να αφήσουμε κατά μέρος κάποιες τροπολογίες. Έχω κάνει μια πρώτη προσπάθεια για συμβαστικές τροπολογίες και θα παρακαλούσα τις ομάδες μέχρι τα τέλη της προσεχούς εβδομάδας να μας ε, δώσουν τα σχόλιά τους. Έχουμε προβλέψει συνεδρία των σκιωδών συγκητών προς τα σαρχάς Νοεμβρίου για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε για τις, σκιώδεις, ε, συμβαστικές τροπολογίες και να καταλήξουμε. Για τον ορίζοντα 2020 λοιπόν έχουμε ε, αναβάλει για τις 20 Νοεμβρίου την έκθεση και γι' αυτό συμφωνώντας και με τον ε, αρμόδιο συγητή είπα να αναβληθεί και η δική μας η πρόταση για τις 20 Νοεμβρίου για την Ολομέλεια. Για τις, μικρο, για τις μικροεπιχειρήσεις που αναφέρονται ρητά προκειμένου να διαφυλαχθεί η ε, συνέπεια στο κείμενο, στη διατύπωση. Προτείνω να ακολουθήσουμε τη διατύπωση του Συμβουλίου και να ισχύει για το κείμενο αυτό ο επίσημος ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που περιλαμβάνει και τις μικρές. Για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επιχειρήσεων. Είμαι διτεθειμένος να δεχθώ μια λιγότερο λεπτομερή ε, ορολογία στο κείμενο με μία απαρίθμηση, αντιθέτω από την προβλεπή μου αρχική τροπολογία και από ό,τι φαίνεται οι βουλευτές συμφωνούν στο σύνολό τους να βελτιωθεί η κάλυψη του δικτύου των επιχειρηματιών. Εγώ σε μια συνάντηση του δικτύου στο Μανχάιμ έμαθα από τους συνομιλητές μου επιχειρηματίε εκεί ότι πολλές φορές είναι πολύ, διαφορε... πολύ μεγάλες διαφορές και ως προς την ποιότητα στο δικτύωση αυτή και άρα χρειάζεται όχι μόνο η τυπική δικτύωση αλλά και η ουσία των ε, πληροφοριών ε, που ανταλλάσσονται και κυρίως θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μεριμνήσει για το θέμα αυτό. Αυτό ισχύει βέβαια και για την ενισχυμένη δικτύωση Γιατί και στη Γερμανία όπου μπορεί να έχουμε τερματικά αυτού του, τερματικές απολύξεις αυτού του δικτύου χρειάζεται καλύτερη δικτύωση μεταξύ των βιομηχανιών, μεταξύ των διαφορών μονάδων ώστε να γνωρίζουν και καλύτερα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το ε, πρόγραμμα. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση του ECR είχε να κάνει με την ε, οικονομική διευκόλυνση του κεφαλαίου διακινδύνευσης και τον περιορισμό της σχετικής υποστήριξης και όσο και αν φαίνεται ενδιαφέρουσα νομίζω ότι θα ήταν πιο σκόπιμο να έχουμε ένα ποσοστό του 30% για να το όριο για να έχουμε περισσότερη ευελιξία στην ε, στήριξη που θα προσφέρουμε. Επίσης, διευκόλυνση έχουμε ένα ποσό περί τα 100.000 ευρώ που ήταν και η πρόταση του Συμβουλίου. Βλέπω ότι είναι πολλοί οι βουλευτέ οι οποίοι θέλουν περισσότερη συμμετοχή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην ε, πρόταση αυτή. Και στρεφόμενος προς την Επιτροπή θα ήθελα να επισημάνω ότι το θέμα δεν είναι να ληφθούν αποφάσεις από την Επιτροπή για τον προσδορισμό των προτεραιοτήτων. Αλλά η πληροφορίες που θα ανταλλαχθούν, η, η γνώση, η εξειδίκευση που θα προσφερθεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις θα βοηθήσει πιστεύω στην καλύτερη κατανομή και των κονδυλίων και την πιο δίκαιη κατανομή. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μου προσφέρθηκε στο στόχο μια, για μια ποιοτική απογραφειοκρατικοποίηση με ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς στόχους που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κύρια προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια η ποιότητα έχει πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα, αλλά όχι πάντα. Πολλές φορές και οι ποσοτικοί στόχοι έχουν νόημα να τεθούν για να επιτύχουμε ένα φιλόδοξο επίπεδο. Για τις ε, τουριστικές επιχειρήσεις τώρα γνωρίζω ότι και η Επιτροπή και πολλοί συνάδελφοι από την Ιταλία και την Ισπανία αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην στόχευση αυτή. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση να στηρίξουμε και τουριστικές επιχειρήσεις. Το έχουμε άλλωστε ε, περιλάβει και στο κείμενο, αλλά διερωτώ με το εξή. Θα πρέπει να αναδείξουμε έναν ιδιαίτερο κλάδο ενώ πρόκειται για μια πρόταση που αφορά όλους τους τομείς και κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και ναι, πιστεύω ότι αν πρόκειται για υπερσυνοριακέ ή διασυνοριακέ δραστηριότητε τουριστικέ, θα πρέπει να ληφθεί ο τουρισμό υπόψη και να στηριχθεί, όπω λέει και η πρόταση τη Επιτροπή. Αλλά όχι, όχι με ιδιαίτερη αναφορά, γιατί υπάρχει και ο χώρο τη κοινωνία πληροφορία και ο χώρο τη καινοτομία ε, και της δημιουργικότητας και εκ τούτου δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε έναν ιδιαίτερο κλάδο. Δεν θα ήθελα να προχωρήσουμε σε αντιπαράθεση, αλλά νομίζω ότι με μια ειδική οδηγία ή καλύτερα κανονισμό που θα στοχεύει στον κλάδο αυτό θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε κύριε Κρότσμαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Μπέντσεν, τον κύριο Κρόιτσμαν για το πνεύμα συνεργασία που έδειξε και την πολύ αξιόλογη έκθεση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή έκθεση και θα ωφελήσει όλε τι ευρωπαϊκέ ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επίση, συμφωνώ με τον κύριο Κρόιτσμαν, τον εισηγητή, ότι όταν μιλούμε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τρία είναι τα βασικά θέματα. Πρόσβαση στι αγορέ, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, νομίζω ότι είναι λογικό να έχουμε ένα στόχο. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις αγορές, θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις με τα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν μέτρα για την διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά. Επίσης, ε, θα πρέπει αυτό το δίκτυο ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να επεκταθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά προς το παρόν και περιμένω τη συζήτηση των τροπολογιών, γιατί πολλές είναι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, αλλά ευελπιστώ ότι η τελική έκθεση θα είναι πολύ θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πατρίτσια Τόγια. Ευχαριστώ και εγώ εν συντομία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες και θα είναι δύσκολο να συνδυάσουμε την ανάγκη να είμαστε περιεκτικοί και σύντομοι με τις πολυάριθμες τροπολογίες που κατατέθηκαν. Πάντως, δυστυχώς δεν έγινε πρώτη συζήτηση με τους κοιόδης συγκητές. Ε, θα εξετάσουμε το θέμα στις ομάδες μας ε, και θα δούμε αν υπάρχουν και άλλοι ε, σκιώδεις που συμφωνούν μαζί μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όπως ε, ακούσαμε το πρωί από τον εισηγητή, γίνεται μία παραπομπή στον ε, ισχύοντα ορισμό. Ίσως όμως θα πρέπει να τον εμπλουτίσουμε κάπως. Γιατί Ζήσαμε αρκετά χρόνια μια οικονομική και βιομηχανική κρίση και είδαμε ότι η κοινωνική οικονομία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί εδώ μιλούμε για πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκτός από τις μικρομεσαίες. Πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι κατά ανάγκη ιδιαίτερα επικερδείς, αλλά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ε, κοινωνικής οικονομίας. Αυτό δεν καλύπτεται από τον υπάρχοντα ορισμό. Επίσης μιλούμε για την ανάγκη καινοτομίας ε, επιτακτική για την ε, σταθερότητα της οικονομίας και την ε, απασχόληση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον τουρισμό με την πληροφορική ή άλλους κλάδους της οικονομίας. Τουρισμός είναι ένας ολόκληρος, μια ολόκληρη βιομηχανία και δεν ενδιαφέρει μόνο ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλες, γιατί παντού υπάρχει προσφορά και ζήτηση για τον τουρισμό. Είναι ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος, λοιπόν, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τέλος, υπάρχουν κάποια προβλήματα δημοσιονομικά. Καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε το κόσμο, το Horizon ή τα διαρθρωτικά ταμεία. Να συνδυάσουμε και να συντονίσουμε τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης ε, για να δρομολογήσουμε τα προγράμματα. Αυτά τα σημεία χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευση και διευκρίνηση, αλλά είμαι πρόθυμη να συνεργαστώ με τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένας τρόπος ε, αποτίμησης της σπουδαιότητας μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι ο αριθμός των ε, τροπολογιών που κατατίθενται. Έχουμε στην περίπτωση αυτή 464 ε, τροπολογίες, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον που προκάλεσε στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό και το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι γνωστή η σημασία του κλάδου αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 98% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και εξασφαλίζουν τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότερες όμως από αυτές δυστυχώς διανύουν μια πολύ δύσκολη στιγμή στα κράτη-μέλη. Στην πατρίδα μου για παράδειγμα, την Ισπανία, γνωρίζω πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ε, πολύ υγιή και εύρωστα χαρτοφυλάκια είναι απόλυτα βιώσιμες, αλλά δυστυχώς ε, ξαναγκάζονται σε κλείσιμο γιατί δεν έχουν ε, δυνατότητα δανειοληψίας από τις τράπεζες. Ε, έχει στεγνώσει η ρευστότητα στην αγορά και αυτό είναι μοιραίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις βιώσιμες με τεχνολογία και ενοτομία που εξαναγκάζονται να κλείσουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο, δεν έχουν πρόσβαση στο δανεισμό. Καλό θα ήταν λοιπόν όχι μόνο να βοηθήσουμε στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά να βοηθήσουμε αυτές που ήδη υπάρχουν, γιατί σε πολλές χώρες μέλη τέτοιες επιχειρήσεις ε, διανύουν χαλεπούς καιρούς. Ελάχιστο, ελάχιστη πρόσβαση σε δανεισμό, υπερβολικό κόστος, γραφειοκρατικό άχθος. Οπότε όλες οι τροπολογίες που στόχο έχουν την ε, άρση των γραφειοκρατικών φραγμών και των διοικητικών διατυπώσεων, τη δημιουργία απλών μεθόδων για τη ε, δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την εξασφάλιση τη ρευστότητα στην αγορά, όλε αυτέ οι τροπολογίε είναι ζωτική σημασία. Και εγώ προσπάθησα με τι δικέ μου τροπολογίε αυτά τα σημεία να υπογραμμίσω. Και όχι μόνο εγώ φυσικά, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ σημαντική αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία και συγχαίρω θερμά τον εισηγητή μα τον κύριο Κρόιτσμαν για το έργο του και ευελπιστώ ότι θα συμβάλλουμε με την πρότασή μας να ανακουφίσουμε κάπως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Μασέσκου Κουκόβιτς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Κρότσμαν. Εξαιρετική έκθεση και απολύτως απαραίτητη στις μέρες μας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περιμένουν κάποιες διευκολύνσεις για να επιβιώσουν στο μέλλον. Περιμένουν την μείωση της γραφειοκρατίας, περιμένουν να δουν δράση. Και αυτό αφορά τόσο τις ε, υφιστάμενες λειτουργούσες εταιρείε όσο και αυτές που ξεκινούν σήμερα. Για όλες αυτές η Θεοκρατία συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο. Για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων είναι προφανές ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρόκειται για ταχυδρομικές στηρίδες. Ε, πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους που περιμένουν τη βοήθειά μας. Αν ε, θέλουμε να διεισδύσουμε σε αγορές και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Πρέπει οι ευρωπαϊκές αυτές επιχειρήσεις να συνδεθούν περισσότερο χάρη στην σύγχρονη τεχνολογία με κέντρα γνώσης και το καθεξής. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω από την Σλοβενία, ότι οι επιχειρηματίες περιμένουν από εμά να κάνουμε κάτι καινούριο και διαφορετικό. Το λόγο έχει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δ. Χέρμπερτ. Καλημέρα σα. Εκ μέρου τη Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν, τον εισηγητή, αλλά και όσου συνέβαλαν στην έκθεση αυτή. Έχετε δίκαιο το κόσμο είναι το μόνο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε ειδικώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και σήμερα είναι ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα τα οποία φύγουν και στις τροπολογίες. Το πρώτο αφορά τους στόχους. Στις τροπολογίες βλέπουμε δύο κατευθύνσεις, δύο γενικές κατευθύνσεις. Ορισμένοι θέλουν να προσδιορίσουν περισσότερες λεπτομέρειες και να θέσουν όρια στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων. Εμείς εν προκειμένου θα λέγαμε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για ένα επταετές πρόγραμμα πλαίσιο, άρα ας αφήσουμε περιθώρια ευελιξίας, ας μην περιορίσουμε υπερβολικά τα περιθώρια δράση μας τα επόμενα 7 χρόνια. Άλλες τροπολογίες που αφορούν και πάλι τον στόχο βαίνουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του στόχου και προκειμένου συμφωνώ με τον εισηγητή ο οποίος μας είπε ότι όσο ευρύτερο είναι ο στόχος με τον ίδιο προπολογισμό τόσο περιορίζεις στην πράξη τη δυνατότητα να κατανείμεις τους πόρους αυτούς με τρόπο αποτελεσματικό. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατηρήση. Δεύτερον, για την μείωση του διοικητικού φόρτου. Εν προκειμένου, συμφωνούμε απολύτω με το Κοινοβούλιο. Δρομολογήσαμε την πρώτη προσπάθεια στον τομέα και πιστεύω ότι θα υπερακοντήσουμε τον στόχο του 20%. Δεν ξέρω πώς θα υπερβούμε όμως αυτό το στάδιο και εκεί οι επιχειρήσεις μας στέλνουν σαφώς το μήνυμα ότι δεν βλέπουν ακόμη το ποιοτικό άλμα που περιμένουν στον τομέα αυτών της μείωσης, δηλαδή της γραφειοκρατίας. Ένα από τα θέματα βεβαίω είναι πώς θα μετρήσουμε την επίτευξη του στόχου. Αλλά από εκεί πέρα το θέμα είναι να εντοπίσουμε τις προσπάθειές μας στα βασικά εμπόδια. Και αυτό εδώ το δεύτερο είναι κρίσιμη σημασίας. Τρίτη παρατήρηση. συνεννόηση και συγκέντρωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εδώ συμφωνούμε απολύτως με το Κοινοβούλιο και ήδη είμαστε σε επαφή με τι οργανώσει που εκπροσωπούν τι μικρομεσαίες. Το παράδειγμα τη μείωση τη γραφειοκρατίας είναι μια τέτοια προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας και το εξή. Μην μας παρακαλώ να συμπεριλάβουμε τις ενώσεις των μικρομεσαίων στην εφαρμογή, στην υλοποίηση του προγράμματος, όπως ζητούν πολλές τοπολογίες... διότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις συμφερόντων, διότι οι ενώσεις αυτές είναι και οι δικαιούχοι των αποτελεσμάτων της προσπάθειας. Ο κ. Κρότσμαν ευτυχώς είπε ότι είναι υπέρ μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, προκειμένου και από αυτού, όπως είπα, συμφωνούμε και εμείς απολύτως. Όσον αφορά το δίκτυο επιχειρήσεων, εννοείται ότι θα τους βοηθήσουμε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και ποιοτικώς πιο αποδοτικοί. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Σε ευχαριστούμε. Θα δώσουμε ξανά το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Κρότσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ναι, και έχει περάσει η ώρα. Νομίζω ότι θα είναι καλό ο κανονισμό στον οποίο θα καταλήξουμε. Το είπα και νωρίτερα ότι θα συναντηθούμε με του σκιώδει ηγητέ την επόμενη εβδομάδα, θα συνεργαστούμε, θα του να βρούμε καλέ συμβιβαστικέ τροπολογίε και να φτιάξουμε έτσι ένα καλό κανονισμό και περιμένω βέβαια και τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. gli ε, emendamenti. Οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν ή μάλλον ε, μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου. Μπορούμε να περάσουμε στις ε, ψηφοφορίες τώρα. Ελπίζω να έχετε φέρει όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες σας. Ας κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι, ποιος είναι υπέρ, μία δοκιμή για το μηχάνημα, άρχεται η ψηφοφορία. Και και κόντρο. Κατά, αποχές. Scusatemi, proviamo a rifare, ho sbagliato anch'io. Allora... Συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Ας κάνουμε, παραλαμβάνω, μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Chiusa la votazione. Τέλος ψηφοφορίας. Ο πίνακας δεν λειτουργεί. Non era il numero, è che non funziona, non funziona il tableau alle nostre spalle. Όχι, ο πίνακας εδώ πίσω δεν λειτουργεί. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έκθεση Κορέιρα Campos. Τροπολογία 188. Θα ψηφίσουμε συνολικά ποιος είναι υπέρ. Μια στιγμή όλα. Είναι παρόν ο εισηγητής Αντώνιο Φερνάντο κοχαίρα Κοχαϊα-Δεκάμπος. Έχουμε την πρώτη μας ψηφοφορία που είναι οι διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Ο εισηγητής μας ε, είναι έτοιμος. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ξεκινούμε λοιπόν από την τροπολογία 188. Ψηφίζουμε συνολικά διάφορες τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της ΕΚΟΝ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της Επιτροπής Περιβάλλοντος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της Επιτροπής Ρέτζι. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 189. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Μόνο δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι λίγο περίπλοκη αυτή η ψηφοφορία, γι' αυτό σας παρακαλώ από τώρα να δείξετε υπομονή. Τροπολογία 205. 205, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 248, δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, τη βρήκατε, υπέρ. Μια στιγμή, μια στιγμή. Σιγά σιγά. Τροπολογία 248 του εισηγητού Φερνάντο Κοχέα Ντεκάμπος. 248 αυτό, αλλά μόνο το δεύτερο τμήμα. Μόνο το δεύτερο τμήμα της 248. Το βρήκατε? Γιατί οι υπόλοιπα έχουν καταπέσει. Έχει απομείνει μόνο αυτό. Το βρήκατε όλοι? Ε, για μας είναι η σελίδα 9, δεν ξέρω σε κάθε κατάλογο τι νούμερο έχει. 248 λοιπόν τροπολογία, δεύτερο τμήμα μόνο. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3, πρώτο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, Η γραμματεία επιβεβαιώνει ότι ψηφίζουμε την τροπολογία, τη συμβιβαστική τροπολογία 3. Το 187 ήταν μέσα στο σύνολο. Συμβαστική τροπολογία 3, πρώτο τμήμα, παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 286, δεύτερο τμήμα, όπως και πριν, είναι η σελίδα 15 για το ΕΛΚ 10 στον άλλο κατάλογο. Τροπολογία 286, δεύτερο τμήμα. Έτοιμοι όλοι. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 324 παρακαλώ. 324. Είμαστε στη σελίδα 18. Τη βρήκατε. Ποιος είναι υπέρ της 324 κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Με ονομαστική ψηφοφορία λέει η πρόεδρο. Το, την τροπολογία 324. Allora, 25 favore. 25 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία 324. Συμβαστική τροπολογία 4 τώρα, πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 357 σελίς 23 για το ΕΛΚ. Το βρήκατε όλοι, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 418 σε 27 του καταλόγου ψηφοφορίας τροπολογία 418 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία συμβαστική 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 434 παρακαλώ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 6 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 446 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 447 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Συμβαστική τροπολογία 13 μαζί με τις τροπολογίες 44 και 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 45 της Οικονομικής Επιτροπής και 46 της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι υπέρ μαζί, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 14, πρώτο τμήμα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Συμβαστική τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, ε, τροπολογία 80, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 622. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44, έμβη, Επέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 623, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 624, ποιος είναι η και 625 γιατί είναι παρόμοιες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 626, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 627 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 628 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 629 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 της Ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 της ίδιας Επιτροπής υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 81 λάθος. 630. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές. Μάλλον εγκρίνεται 630, αλλά ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 630 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Περισσεύει μία ψήφος του ΕΛΚ. Τέλος ψηφοφορίας 28 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται 630. Συμβαστική τροπολογία 16. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 670. Περνάμε στην 670. Του Γκαστόν Φράγκο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 670 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Και περνάμε στην 84. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον απορρίπτεται. έχει ήδη καλυφθεί. Συμβαστική τροπολογία 17, πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 692, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 692 άρχιτη ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 692 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. 26 υπέρ 28 κατά, απορρίπτεται 692 και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 18, πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ? Κατά, αποχές, εγκρίνεται. «724. Ποιος είναι υπέρ» «Κατά» Μάλλον εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 35 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 τώρα. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 763. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 790. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 117. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 120. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της Ρέγγι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της Τραν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 της Ρέτζι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 121 για την αιτιολογική σκέψη 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 122. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 122 λέει πρόεδρος, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 Συνήθως θα συμφωνούν οι δύο μεγάλες ομάδες, ισχύει αυτός ο κανόνας. Θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αλλά θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 122, πολύ ευχαρίστως. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 25 υπέρ 29 κατά. Απορρίπτεται. 123. A favore. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 123. Τέλος ψηφοφορίας. 29 κατά, άρα απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 124. Τέλος. 31 υπέρ 22 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της ΕΚΟΝ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 έμβη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 Ρέτζι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα. Γιατί αν δεν ψηφίζετε όλοι, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 25 προς 27. Τροπολογία 125. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμβη. 2. Υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2 της ΕΜΒΗ. Αλλάζουν οι συσχετισμοί. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 22 προς 32. Πάμε στην τροπολογία 4 της περιφερειακής. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 129. Παρακαλώ όταν έχουμε οριακό αποτέλεσμα να ψηφίζουν τα μικρότερα κόμματα γιατί δεν βλέπουμε αν εγκρίνεται ή αν 31 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται 129. Τροπολογία 3 της Έμβη και 5 της ΡΕΤΖΙ υπέρ, είναι ταυτόσιμες γιατί η τροπολογία 2 της ΣΥΜΚΟ έχει καταπέσει. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τη 2. Την 3 και την 5, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η 130. Τροπολογία 3 της τράν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 131 μαζί με την τροπολογία 4 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 μαζί με την τροπολογία 2 της ΕΚΟΝ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 136 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 138 παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 23 προς 27 ψήφι. Απορρίπτεται λοιπόν 138. Τροπολογία 6 της Ρέγγι. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 του συγκεκριτού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141. 141 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ ή μάλλον λάθος λέει η μαλλον λαθος λεει ο προεδρος 144 4, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ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 εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 152. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 157 άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας 30 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται Τροπολογία 8 τη επιτροπή Μεταφορών υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 158, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 9 τη Ρέγγι υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 τη επιτροπή Τράν υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 10 τη επιτροπή Μεταφορών υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 161 υπέρ ε, με την 4 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 162 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 της έμβι. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της ΡΕΓΚΙ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 της Επιτροπής Μεταφορών, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της εκών. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 της ΡΕΓΚΙ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία οι τέσσερα καταπίπτουν οι υπόλοιπες. Πάμε στη 12. Ποιος είναι υπέρ κατά της Επιτροπής Μεταφορών. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ρέτζι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 της Στράν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 έμβη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 της ρέγγι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 της τράν υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 15 της Επιτροπής Μεταφορών. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 30 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 171. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Ήμκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175 και 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 7 του εισηγητού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 και 6 της εκών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 179 και 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται απορρίπτεται. 16 τη επιτροπή Μεταφορών υπέρ, κατά, απόχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 8 του εισηγητού υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Από την 182 ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 17 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 εκών. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 8 εκών, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τα θεωρώντας 115 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για τις τροπολογίες. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Allora, 49 a και 1 contrario contrario, 49 υπέρ, μία ψήφος κατά 6 αποχές. Τώρα, ψηφίζουμε για τις διαπραγματεύσεις, ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Λαμπρά, 55 υπέρ, μία αποχή μόνο για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια Κύριε Κορέα Κάμπος, έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ψηφοφορία, για την ιόβια υπομονή που έδειξαν οι συνάδελφοι με αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη λίστα της ψηφοφορίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους και οδησηγητές και όσους ε, συνέβαλαν στην κατάρτιση της έκθεσης. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και πολύ ενεργό στη συμμετοχή τους. Και επίσης ε, να αναφέρω ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια και της Προεδρίας Επιτροπής για τις ε, διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουν. Έχουμε το το Υπουργικό Συμβούλιο Ενέργειας στη Λευκοσία και Υπάρχει πρόθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής και θα ήθελα και εμείς να υποστηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία να διεκπαιρεωθεί η νομοθετική διαδικασία για το σημείο αυτό μέχρι τα τέλη του έτους. Ελπίζω να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Οπότε περνάμε... Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Λιγότερο περίπλοκη από την προηγούμενη, αλλά πάντως αρκετά γεμάτη. Γι' αυτό θα σας δείσω να δείξετε και άλλη υπομονή αφού είναι κάπως δύσκολο οπότε, να διαγνώσουμε τα αποτελέσματα. Ξεκινούμε με την έκθεση του κυρίου Ρίουμπιχ, λοιπόν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 μαζί με 45 τροπολογία υπέρ κατά έχει αποσυρθεί έχει αποσυρθεί ζητά ο συγγνώμη λέει πρόεδρος και εμείς κάνουμε λάθη 25, τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά άποχες. Δεν το βλέπω καθαρά. Επαληθεύουμε. Πέρασε τις ε, ψηφοφορίες. 25 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υ... όχι. 37. 37 λέει πρόεδρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει η 53 πάμε στην 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8β συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρώ στην παράγραφο 12, προφορική τροπολογία του εισηγητού, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρώ σε μια ομού ψηφοφορία των 62, 64, 65, 66 και 67 τροπολογιών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. «Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 91 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Μάλιστα. Την 91, επαληθεύουμε την υπαριθμόνα 91 τροπολογία με προφορική τροπολογία. Πέρα στις ψηφορίες. 17 υπέρ. 36 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχή. Να το επαληθεύσουμε, λέτε. Όχι, εγκρίνεται λοιπόν. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 102 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 104 και 105 έχουν καταπέσει και πάμε στην 107. Λοιπόν υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε την 107 τροπολογία. 107. 107. Πέρα στις ψηφοφορίες. Τριάντα υπέρ 24 κατά εγκρίνεται.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 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 133 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 147 και 146 και 148 όχι, όχι μόνη της 147 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 146 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ας κάνουμε μια παλήθευση αν θέλετε για την κυρία Τόγια πέρασε τις προφορίες. 14 υπέρ 39 κατά απερίφθη 148 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στις αιτιολογικές προτάσεις, πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αιτιολογικές σκέψεις 3, τροπολογία 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται.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 Και τώρα έχουμε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου την, ε, τη γνωμοδότηση 3, η τρίτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 8 της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 της ΣΥΝΤΑ υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10, ε, λέει πρόεδρος υπέρ κατά 18 και 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 της απασχόλησης υπέρ έμπλο όχι δεν ψηφίζεται στην απασχόληση τώρα πάμε Ε, είναι λάθος το φίλο που μου δώσατε λοιπόν. Δε, δύο της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τέσσερα της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα της απασχόλησης υπέρ Κατά. Όχι, η 7 πρώτα. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά απόχέ. Δεν ψήφισε κανεί τίποτα. Ούτε υπέρ ούτε κατά. 14 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα αλλάζουμε σελίδα και πάμε στη 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ όχι όχι όχι 21. Όχι, καταπίπτει 21. Πάμε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. 1, 2, ε, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 5, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 6, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 8 της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 10 της Ρέτζη, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 11 της Ρέτζη, υπέρ, κατά,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 κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Α, ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές και συγχαρητήρια στον κύριο Ρεπίχ. Τώρα περνάμε στην έκθεση του κύριου Κόβατς. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά αποχές. Απερίφθη. Πέντε υπέρ. Όχι, στο 5 λοιπόν πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Φαίνεται να έχει απορριφθεί. Ας επαληθεύσουμε. Την 5 υπαριθμών 5 τροπολογία. Πρώτο τμήμα. Πέρασε τη προφορία. 28 υπέρ, 28 κατά. Απερίφθη. Δύσκολη ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ίδιε ισορροπίες βλέπω να εκφράζονται. Ας επαληθεύσουμε λοιπόν. Πέρασε. 24 υπέρ. Και κατά. Απερίφθη λοιπόν. Πιο ψηφίσει ισορροπίε. Ε, τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Απερίφθη. 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τελική ψηφοφορία για τις τροπολογίες ηλεκτρονική παρακαλώ Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 51 υπέρ, 4 αποχές. Καμία ψηφος κατά. Για τις διαπραγματεύσεις, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 55 υπέρ. Πολύ καλό. Μπράβο σας, συγχαρητήρια στον συνάδελφο κύριο Μπέλα Κόβατς. Και έχουμε μία ψηφοφορία μόνο για το νομοθετικό ψήφισμα, σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, μία ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον κύριο Κόβατς πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. πέντε υπέρ, μία εποχή. Και τώρα πάμε στην έκθεση κυρία Τζαβέλα. Τροπολογία 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 32 υπέρ 24 κατά. Εγκρίνεται. Λάθος έκανα. Συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 33, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την 35 Έχουμε μία προφορική τροπολογία αλλά η κυρία Τσικάου δεν συμφωνεί με αυτήν και έτσι δεν μπορούμε να δεχτούμε την προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 35 χωρίς την προφορική προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Κιούζα. Τέλος ψηφοφορίας. 35 κατά, απορρίπτεται 35. Τροπολογία 37, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Συμβαστική τροπολογία 5, ηλεκτρονικός έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 31 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 71 παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ και 13 κατά. 71 λοιπόν εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70... Για την 73 επαναλαμβάνει την ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος διορθώνει η πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 27 προς 26 οριακά εγκρίνεται. σε 74 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 80, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 και 105 μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 108 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 και 121 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 125 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άλλαξαν οι αναλογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Περισσεύει μια ψήφος του ΕΛΚ. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 21 ψήφους υπέρ και 31 κατά 122 τώρα. ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ναι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απορρίπτεται, λέει πρόεδρος. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 177 προηγουμένως. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, ψηφοφορία 43 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται 177. Συμβαστική τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 182 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 ή μάλλον 206 διορθώνει η πρόεδρος του κυρίου Μπιούτι Κόφερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε 208, 9, 10, 11 και, 11, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές. Μάλλον εγκρίνονται αυτές τις τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες. Ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνονται όντως 30 υπέρ, 26 κατά. 212 τώρα, ή μάλλον 215 λέει η πρόεδρος, λεει κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 216, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τώρα για τα θεωρώντα, τροπολογία 1 και 2 μαζί, Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχέ. Εγκρίνονται 3 υπέρ, κατά αποχέ. Εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά αποχέ. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ και 23 κατά. Μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε στην έκθεση Μαρινέσκου τώρα. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 μεταφορές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 117 με την 14 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 μαζί με τη 16 Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται απορρίπτεται, τροπολογία 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 125, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 126 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 127 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 14 της Επιτροπής Προπολογισμών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 ναι. υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 132 με τη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 ε, των προπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 με τη 17 των προπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 56, 58, 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 αφέτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155 63 μάλλον. 63 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 μεταφορές υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 μεταφορές υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 μεταφορές υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67, 68 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73, Α, το κάναμε. 69, 69 ε, υπέρ, τροπολογία 69 του εισηγητού. Υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15, υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 173 και 30 των μεταφορών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά αποχές μαζί με την 34 των μεταφορών, κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 του εισηγητού. 76. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 77 και 36 μαζί. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνονται. 182 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 183 και 184 μαζί υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνονται. 23 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 189 και 22 των προπολογισμών υπέρ. Κατά απόχε εγκρίνονται. 21 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 191 και 39 τη τραν μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά αποχές εγ, απορρίπτεται. 192 υπέρ κατά «192 υπέρ» κατά αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται. Αφέτ 1. Υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αφέτ, υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αφέτ, υπέρ, κατά απόχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Προπολογισμοί υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Αφέτ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 αφέτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 αφέτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της Τραν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 της Αφέτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της ΑΦΕΤ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 των προπολογισμών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 μαζί με την 8 των προϋπολογισμών. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 7 των μεταφορών υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 31, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 του συγητού, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 13 της αφέτη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 της ΑΦΕΤ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 των προπολογισμών, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 της ΑΦΕΤ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 17 της ΑΦΕΤ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 110, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 των προπολογισμών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται παρακαλώ η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 49 ψήφισαν υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις εντολή άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας 53 υπέρ. Πανψηφί εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες μας. Βλέπετε, σήμερα τελειώσαμε πολύ νωρίτερα, ενώ χθες δεν προλαβαίναμε να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Βιντάλ Κουάδρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο παρατηρήσεις μόνο. Πρώτον, να σα συγχαρώ θερμά για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγατε αυτή την ε, μακροσκελή ψηφοφορία και μάλιστα την ολοκληρώσετε και με ταχύ ρυθμούς. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Δεύτερο σχόλιο. Όσοι έχουμε κάποια εμπειρία ως ηγητές και όδης ηγητές, γνωρίζουμε ότι πολλές φορές, ότι, πολλές φορές ο αριθμός των τροπολογιών εξαρτάται από τις προσπάθειες του εισηγητού και των σχεδόν εισηγητών να καταλήξουν σε, διαπρα... σε συμβαστικές προτάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ενδύνουμε αυτές τις προσπάθειες και να τις εξάρουμε. Γιατί μερικές φορές το συνεργάσιμο πνεύμα μας οδηγεί σε καλύτερες και περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες ώστε να περικόπτουμε σε τελική ανάλυση τον χρόνο των ψηφοφοριών και να αποφεύγουμε τέτοιες μακροχρόνιες ψηφοφορίες. Εντάξει, ολοκληρώσαμε. Ραντεβού τώρα στις 3. Διακοπή προς το παρόν. Γεια σας.